ψηφοφορία αύριο στις 12 το μεσημέρι. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης κοινή συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας και το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης οι εκθέσεις Μέλο και Λάντφορντ. Θα δώσω τον λόγο στους ηγητές. Ξεκινάμε με τον κύριο Μέλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η έγκριση αυτής της οδηγίας σημαίνει ε, του εγκλήματος και ενός μέσου έρευνας. Το Σέγγεν ήταν θεμελιώδες στην οικοδόμηση αυτή, αλλά η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εμπορευμάτων υπηρεσιών και κεφαλαίων επέτρεψε ε, ακόμα περισσότερα εγκλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να τα καταπολεμήσουμε, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διασυνοριακό έγκλημα που δημιουργεί μεγάλους ε, κλειδονισμούς, διαφθορά, ε, τρομοκρατία, εγκληματικές πράξεις σε διασυνοριακή βάση. Στη περίπτωση Μέρλιν Μακέιν ξέρετε ότι ε, συμμετείχαν δύο χώρες, η Πορτογαλία και το Ενωμένο Βασίλειο και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία στο μέλλον. Η οδηγία δεν αλλάζει την τήρηση των δικαιωμάτων και τις νομικές αρχές που αφορούν το έκτο τμήμα της συνθήκης. Αλλά η απόφαση για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας θα βοηθήσει το κράτος έκδοσης έτσι ώστε να εκδώσει αυτή την εντολή και στη συνέχεια μετά από την διαδικασία ανάκρισης και συλλογή αποδείξεων να μπορέσει να εφαρμοστεί στη χώρα ε, υποδοχής. Θα πρέπει να συλλέξουμε στοιχεία DNA, πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς ή χρηματοοικονομικές κινήσεις, κάτι το οποίο θα συζητηθεί μεταξύ των δύο κρατών και θα υπάρχει τυποποίηση αυτών των στοιχείων από την οδηγία αυτή. Επίσης θα πρέπει να τηρήσουμε το κράτος δικαίου και να υπάρχει σωστό καθεστώς υπεράσπισης. θα πρέπει να υπάρχει, να προστατεύεται και το δικαίωμα προσφυγής. Αυτή η διοικητική απλούστευση και η μείωση της γραφειοκρατίας θα πρέπει να οδηγήσουν στην καλύτερη διάρθρωση και συνεργασία στη πλαίσια της διερεύνησης εγκλημάτων. Πρόκειται για πολυσχηδείς διαβουλεύσεις που είναι μακροχρόνιες πολλές φορές και έτσι δεν φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και ανέκυψε και αυτή η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις διάφορες προεδρίες από την Δανέζικη ε, μέχρι την Ιρλανδική ε, και την ελληνική και τον κύριο Βάισεν Χόλερ, την κυρία Λάτφορτ, τον κύριο Τίμωθη Κίρκοπ ε, και τον κύριο Ντεάν, διότι μας βοήθησαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Η Βαρόνι Λάντφορτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έγκριση της έκθεσής μου για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης νομίζω θα συνεισφέρει στην Ευρωπαϊ... στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Όπως και ο κύριος Μέλλο θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδελφούς για τον υψηλό βαθμό συνένεσης για τις νομοθετικές αλλαγές. Όλες οι πολιτικές ομάδες που συμμετείχαν στις ε, συνεδριές των σχεδόν συγητών μας στηρίζουν πλήρως. Επίσης μας βοήθησε και η μονάδα Ευρωπαϊκής Προστομής Αξίας της Γραμματείας και η εξαιρετική ε, έρευνα των καθηγητών Βέμπερ και Αλέντιου με τους οποίους ευχαριστώ. Βλέπουμε πως οι αρχές αντιμετωπίζουν συχνά περίπλοκα διασυνοριακά εγκλήματα και πρέπει να κρατήσουν τους πολίτες ασφαλείς. Το υποστήριζα αυτό ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο χιλιάδες καταδικασμένοι εγκληματίες ε, εκδίδονται πάρα πολύ πιο γρήγορα από τις παραδοσιακές διαδικασίες οι οποίες εμπλέκουν υπουργού. Εξάλλου μην ξεχνάμε πως όταν η δικαιοσύνη καθυστερεί δεν είναι πλέον δικαιοσύνη. και βεβαίως η όλη υπόθεση είχε ξεκινήσει από το Συμβούλιο Ιστορικών και Δικαιοσύνης αλλά χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις καθώς είχαν αγνοηθεί οι ευρωβουλευτές. Οπότε υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές και πρακτικές και άρα σωστά ασκήθηκε κριτική πως πρέπει να βελτιωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ήταν σωστή αυτή η κριτική και όχι η ιδεολογική κριτική η οποία ασκήθηκε. Επίσης, η ad hoc και ασυντόνιστη δράση δεν είναι βεβαίως ο κατάλληλος τρόπος συνεργασίας για να επιτρέψει σε σώματα ασφαλείας, εισαγγελείς, δικαστήρια να ξέρουν ποιες είναι οι διαδικασίες και τα δικαιώματα και Μόνο λοιπόν ένα ενιαίο πλαίσιο θα είναι εγγύηση αποτελεσματικής άσκησης της δικαιοσύνης σεβόμενο τα θεμελιώδη δικαιώματα των κατηγορουμένων. Έχουμε λοιπόν ένα έτος μπροστά μας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αν επανεκλεγώ θα συνεχίσω να πιέζω. Θα πρέπει βεβαίω να δούμε και την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας καθώς συμπληρώνει το ένταλμα σύλληψης και ασκεί πίεση και νομίζω πως δημιουργεί ένα προηγούμενο. Το πρώτο είναι ο έλεγχος αναλογικότητας, καθώς η εκδούσα αρχή πρέπει να δει εάν είναι πραγματικά αναλογικό το ένταλμα και δεύτερον βεβαίως υπάρχει η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έκθεσή μου προτείνει αυτά να μεταφερθούν και στο ένταλμα σύλληψης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει και η ανταλλαγή πληροφοριών, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε πω το Ευρωπαϊκό Τέλμα Σύλληψη δεν θα χρησιμοποιείται για να ρίχνουν άδεια και να φτιάνουν γεμάτα οι αρχέ, για να τσιμπάνε υπόπτους και όχι πραγματικά ανθρώπους οποίους θα ασκηθεί δίωξη. Τα άτομα δεν πρέπει επίσης να περνάνε υπερβολικά μεγάλο χρόνο σε προφυλάκηση ενώ προετοιμάζεται η εισαγγελία. Θα πρέπει επίσης η Ευρωπαϊκή Έντολη ε, Έρευνας να αφαιρέσει κάποιο από τον φόρτο του εντάλματος σύλληψης. Τα υπόλοιπα θα τα, θα καλύψω, με συγχωρείτε, στη δευτερολογία μου. Αλλά αναμένω και την απάντηση της ε, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο και την Πρόεδρος Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί κύριοι βουλευτέ, πρώτα από το την μέλου. μέλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη προσεκτικά τη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά την λόγω πρωτοβουλία των κρατών μελών σε σχέση με αυτήν την εντολή έρευνα στις ποινικέ υποθέσεις. Θα μπορούσε αυτή η οδηγία να είναι ένα εργαλείο να κατανοήσουμε το διεσυνορικό έγκλημα και μπορεί να μας βοηθήσει να προσάγουμε στην δικαιοσύνη του φέρουμε ω εγκληματίε. Θα πρέπει όμω να εφαρμοστεί σωστά, να χρησιμοποιηθεί σωστά. Έτσι θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τη σύμβαση για την δικαστική συνδρομή και επίσης ε, την απόφαση ε, ε, τη σχετική με τις αποδείξει. Ε, αυτά ξεκίνησαν το 2008 και έχουν εφαρμοστεί μόνο από δύο κράτη-μέλη. Ελπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα έχουν άλλος, γιατί προσδοκούμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία ορθά και έγκαιρα και για αυτόν τον τρόπο να μην μείνει νεκρό γράμμα ακριβώ όπως έγινε με το ευρωπαϊκό ένταλμα το σχετικό με τις ε, αποδείξεις. Θέλουμε τώρα να καλύψουμε αυτές τις τρεις οδηγίες, αυτές που είχαν προηγηθεί του, ε, της Λισαβόνα. της Λισαβόνας όσον αφορά ε, την, αναστολή και, και άλλες, ε, άλλα εντάλματα εκτός της σύλληψης. Οπότε, Έτσι θα ισχύσει το κοινό χώρο δικαιοσύνη. Βέβαια, έχουν ήδη εκπνεύσει οι προθεσμίε υλοποίηση. Δεν έχουν μεταφέρει τα μισά κρατημέλη τι εν λόγω αποφάσει. Ε, τι έχουν μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο. Θέλουμε έναν χώρο ασφάλεια, δικαιοσύνη και λοιπόν όπω ορίζει το, το άρθρο 3 τη συνθήκη. Αυτό μπορεί το πετύχουμε μόνο εάν τα κράτη-μέλη ε, σωστά υλοποιούν ε, αυτά επί των οποίων έχουν συμφωνήσει. Θέλω να εισηγήσω τον κύριο Νόνο, να τον κύριο Μέλο, τον εισηγητή, αλλά και τους κύριους διότι επιτέλους ένα έργο αξιόλογο. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χαιρετίζει το, το, το κείμενο του κύριου Μέλο και επίσης ότι θέλει να αναβαθμίσει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό θα βοηθήσει πολύ και για άλλη μια φορά τονίζουμε το πόσο σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία της συναποφάσεως. Τώρα, επί της ε, έκθεσης Λατβόντα. Έγινε πρόσφατα συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και σε άλλες ε, περιστάσεις εγώ κατηγορηματικά υπερασπίστηκα το δικαίωμα των Ευρωπαίων για την ελευθερία διακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ανοιχτά σύνορα δεν σημαίνουν ότι οι εγκληματίες μπορούν να διαφύγουν τις δικαιοσύνες απλώς πηγαίνοντας σε άλλο κράτος μας. Και γι' αυτό και χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Ξεκινήσαμε το 2004 αυτή τη διαδρομή. Είναι αποτελεσματικό μέσο ούτω ώστε να συλλαμβάνονται κάποιοι οι οποίοι είναι υποπτή για κάποιο έγκλημα σε άλλη χώρα. Να μην κρύβονται οι καταδικαστέντες ε, σε αυτόν τον χώρο δικαιοσύνης. Έχουμε πάρα πολλά δικαιώματα. Λαθρέμορους, ε, ε, κάποιους που έχουν διαπράξει ε, σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων και πετύχαμε την προσαγωγή στη δικαιοσύνη σε χρόνο πολύ πιο σύντομο από ό,τι παλαιότερα. Αλλά τώρα έχουμε ακόμη και ύποπτους τρομοκράτες οι οποίοι και αυτοί προσαγωγούνται στη δικαιοσύνη ε, εκεί όπου το. Νομίζω ότι το ένταλμα σύλληψης είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιδέχεται βελτίωση και το ότι δεν μπορούμε να το, το, το κάνουμε καλύτερο. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 στην έκθεση για την εφαρμογή είχε πει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Φερρυπίν, να μην ε, ισχύει το έντελμα σύλληψης για ελαφρά Το Ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα σε σχέση με το έντελμα σύλληψης. Ευχαριστώ την Επιτροπή Λίμπε αλλά και την ε, Σάρα ΛΑΝΤΦΟΡΝΤ. σε ευχαριστώ για την εμπειρογνωμοσύνη τους που βοήθησε σε αυτή την έκθεση και έχουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία καλύπτει η έκθεση. Όλα αυτά πρόκειται να βοηθήσουν το διαρκές έργο μας για να βελτιώσουμε το ευρωπαϊκό σύστημα ε, εντάλματος. Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα πρέπει το έργο των, το, συγγνώμη, η θέση των κατηγορουμένων να κατοχυρωθεί, να έχουν δικαίωμα σε διερμηνέα, μεταφραστή, προσβασιμότητα σε συνήγορο για του κατηγορημένου του εναγωμένου. Αυτά θα πρέπει να είναι το ελάχιστο στάνταρ που να ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δυστυχώ κάποια κρατημέρια δεν θέλουν να συμμετάσχουν ε, σε αυτή την πλατφόρμα των ελαχίστων δικαιωμάτων που θα πρέπει να είναι πανενωσιακή. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο τρέχουμε ένα αντίβαρο. Ε, αυτά τα δικαιώματα είναι το αντίβαρο στο ένταλμα σύλληψη. Α πούμε, κάποιοι οι οποίοι συλλαμβάνονται βάσει αυτού του εντάλματο θα έχουν δικαίωμα σε συνήγορο. Αν τα κρατημέλη όμως τώρα δεν ε, ε, εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες, αυτοί που συλλαμβάνουν με το ένταλμα δεν θα έχουν αυτό το δικαίωμα. Οπότε θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν αυτά τα δικαιώματα. Το κοινοβούλιο είναι μια ατομομηχανία. Ε, είναι το κλειδί, ούτως ώστε να πιάσουν τόπο αυτές οι οδηγίε για τα δικονομικά δικαιώματα και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό. Ευχαριστούμε για το ότι πώς βοηθάσατε για τα δικονομικά δικαιώματα για τους ανηλίκους, για τους υπόπτους. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την προσπάθειά μας για τη δικονομία και αυτό θα είναι ένα συμπλήρωμα ιδιώδες ή στην προσπάθεια για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Θα πρέπει όμω όλα αυτά να τα αναδειχθούν όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει ό,τι και να και και υπάρχουν για τα δικαιώματα σε μια δίκη δίκη να κλείσουν, να αρθούν. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, στην έκθεσή σα. σωστά αυτό το ένταλμα σύλληψη ε, μπαίνει στο ευρύτερο πλαίσιο των ε, ε, εργαλείων αμοιβαίας αναγνώρισης, ε, την αναστολή, ε, για την εποπτεία και θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν όλα αυτά πλήρως μεταφερθεί στο ιστορικό των κρατών μελών. Άρα χρειάζεται να δούμε ότι ένα ανοιχτό έντελμα σύλληψη ακόμα δεν μπορεί να πιάσει τόπο, δεν υπάρχουν συνθήκες. Χρειάζεται πρώτα να έχουμε τα, την πλήρη εφαρμογή των ε, ε, αποφάσεων για την αμοιβαία αναγνώση των αποφάσεων. Όταν γίνει αυτό, το οποίο θα είναι το Δεκέμβριο ενός τότε, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε την πλήρη ε, υλοποίηση, εφαρμογή του εντάλματος. Την διαταγή εποπτείας για επίσης και για τις διατάξεις που αφορούν την προσωρινή κράτηση. Έχουμε ε, δίκτυα που προβλέπονται για το ένταλμα σύλληψης. Αυτά ήδη μελετώνται, έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται, είναι πολύ σωστό. Θα συνεχίσουμε προσπαθίες μας. Συμφωνούμε επίσης για το πόσο σημαντικά είναι τα δεδομένα τα αξιόπιστα. Προβάλαμε αυτό το καινούργιο ερωτηματολόγιο για τα δεδομένα που αφορούν το έντελμα σύλληψης. Οπότε όλα αυτά τα οποία έχετε προτείνει πρόκειται να ταιριάξουν το σύστημα του εντάλματος σύλληψης. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρο στον κύριο Κοέλιο Κάρλος. Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, ε, μιλώ εξ ονόματος του ΕΛΚΟΥ και η κυρία Κίνγκαγκέλ δυστυχώς έπρεπε να φύγει από το Στρασβούργο νωρίτερα. Δεν ε, μπορέσαμε να έχουμε μία αξιόπιστη δικαιοσύνη που να είναι αποτελεσματική και αμερόλεπτη, που να λειτουργεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Η ε, ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ σημαντική για να καταπολεμηθεί το διασυνοριακό έγκλημα και να μην μπορέσει κανείς να διαφύγει από τη δικαιοσύνη. Η ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να ε, ανταποκριθούμε, διότι μιλάμε για έναν πυλώνα αμοιβαίας αναγνώρισης από όλες τις δικαστικές αρχές. Πρόκειται για μία νέα πρόκληση, διότι πολλές φορές δεν είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί. Υπάρχουν πολλά χάσματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσα στα πλαίσια αυτού του κατακαιρματισμού της δικαιοσύνης ανά κράτος μέλος και θεωρώ ότι δεν, δεν υπάρχουν έχουν ε, σωστές επαρκείς εγγυήσεις και προστασία του πολίτη. Έτσι δεν υπάρχει πάντα αμοιβαία εμπιστοσύνη. Πολλές φορές δεν γίνονται οι σωστές ε, έρευνες ή επαληθεύσεις. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Λάντφορτ που μιλάει για ελάχιστες προδιαγραφές μέσα στα πλαίσια ε, μίας διασυνοριακής εφαρμογής του ένδικου αυτού μέσου έτσι ώστε να υπάρχει ε, μια καλύτερη ισορροπία διευρωπαϊκά. Η κυρία Λάντφορτ πάντα ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω να αποτελέσει παράδειγμα για τη χώρα της που έκανε opt-out από τον χώρο αυτό των ελευθεριών και της δικαιοσύνης. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον κύριο Νούνο Μέλου γιατί με αυτή του την εργασία φτάσαμε σε μία συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και μπορέσαμε να ε, ανταποκριθούμε εξ αρχής έτσι. Θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ε, και το ένταλμα και την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας μέσα στα πλαίσια αυτού του πακέτου και χαίρομαι διότι ε, λήφθησαν υπόψη τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα και η αρχή του «ne bis in idem». Θεωρώ ότι μπορούμε διασυνοριακά να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα μέσα στα πλαίσια της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων που είναι μία ε, διαδικασία που μέχρι τώρα ήταν αρκετά κατακερματισμένη. Ελπίζω η κυρία Ρέντινγκ να λάβει υπόψη αυτό το διαδικαστικό πλαίσιο και να μπορεί να προβάλλει κυρώσει στα κράτη-μέλη που δεν τηρούν αυτό το πλαίσιο λειτουργίας. Σας ευχαριστώ κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ. Με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ε, θα πρέπει να εκδίδονται πιο γρήγορα και να οδηγούνται ενώπιον του δικαστηρίου ή ε, Όμως ε, καλό αυτό θεωρία, αλλά πάντα υπάρχουν προβλήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δέκα μήνες φυλάκιση είναι η ποινή που απειλεί μία μητέρα ε, η οποία εκδόθηκε από την Πολωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο και ποιος ήταν, ε, ποιο ήταν το έγκλημα της ε, ότι 17 χρονών είχε στην κατοχή της μια μικρή ποσότητα αμφεταμίνης και της είχε επιβληθεί μια ποινή επιτήρησης 10 μηνών την οποία όμως δεν είχε δηλώσει στις αρχές της δεύτερης χώρας στην οποία πήγε το εξακρίβωσαν μόνες της και εδώ πέρα βλέπουμε ποια προβλήματα δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα καθώς η γυναίκα αυτή κινδυνεύει να χάσει την δουλειά της. Εμπιστοσύνη λοιπόν στο σύστημα της δικαιοσύνης ε, απαιτεί να υπάρχει και σεβασμός των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Γι' αυτό ζητάμε από την Κομισιόν να καταθέσει εντός ενός έτους μια νομοθετική πρόταση για τη μεταρρύθμιση του εντάλματος σύλληψης. Κάποια πράγματα. Σε κάθε περίπτωση προέκδοσης του εντάλματος σύλληψης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το βάρος του αδικήματος καθώς και να αναζητά η εκδούσα αρχή μια εναλλακτική λύση. Εάν Επίσης υπάρχει πρόβλημα με τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει η χώρα να μπορεί να αρνείται την έκδοση και οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν. Επίσης χρειάζεται καλύτερος ορισμός των αδικημάτων και δικαίωμα σε δίκαιη δίκη θα πρέπει να υπάρξουν πανευρωπαϊκές ελάχιστες προδιαγραφές όπως το δικαίωμα σε δικηγόρο και διερμηνέα που θα πρέπει να ισχύουν και για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Λάθη παρόλα αυτά μπορούν να συμβούν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ξεκάθαρους κανόνες και επίσης όσον αφορά και την εντολή έρευνας. Οι σοσιαλδημοκράτες δεν αμφισβητούν το μέσο του εντάλματος σύλληψης, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστούν τα πράγματα όπως έχουν μέχρι στιγμής. Γι' αυτό υποστηρίζουμε πλήρως την συνάδελφο την κυρία Λατφορτή. Η Κομισιόν πρέπει να καταθέσει μια νομοθετική πρόταση για να λύσει τα προβλήματα. Και τελευταίο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και στον τομέα του ποινικού δικαίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι πράσινοι υποστηρίζουν την πρόταση αυτή. Μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση όταν κάποιος ζητά, ε, όταν κάποιον αναζητούν οι αρχές μόνο για ανάκριση και όχι λόγω μιας καταδίκης. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιείται το μέσο το οποίο είναι το λιγότερο παρεμβατικό. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει μία ε, εμπιστοσύνη. Εμείς ζητάμε ως πράσινη να υπάρχει ένας έλεγχος αναλογικότητας και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι καλή, αλλά ο έλεγχος είναι ακόμη καλύτερος. Και βεβαίως, όπως λέμε, υγιείστε δια του παραδείγματος. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να αρνηθούμε και την εκτέλεση του ευρωπαϊκού ένταλμα σύλληψης. Καθώς τα τελευταία χρόνια είχαμε πάρα πολύ μεγάλη δυστυχία που προκλήθηκε σε Ευρωπαίους πολίτες με εντάλματα σύλληψης τα οποία εκδόθηκαν με απίστευτη προχειρότητα και οδήγησαν σε προφυλάκηση υποφρικτές συνθήκες. Και το έχω πει επανειλημμένο στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο και η απάντηση που μου έδωσαν ήταν αυτά, τι είναι αυτά, παράπλευρες απώλειες. Μα πείτε τα αυτά σε κάποιον ο οποίος κάθεται προφυλακισμένος και χάνει το σπίτι και τη δουλειά του και τις σχέσεις του. Και τώρα μας λέει η κυρία Ρέντινγκ πως θα αναβάλει τις αλλαγές. Όχι, πρέπει να δείτε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Υπάρχει τώρα 10 χρόνια το Ευρωπαϊκό Σύλληψης χωρίς να υπάρχει όπως είπαμε, το τεστ της αναλογικότητας και να λαμβάνεται απόψη οι φρικτές συνθήκες σε κάποιες χώρες. Θα θέλαμε να λειτουργεί εξίσου καλά παντού, αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και δεν είναι η σωστή βασή για δικαστική συνεργασία. Το ξαναείπα. Καλός ο έλεγχος, καλύτερη η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό εγώ είμαι ικανοποιημένη με την έκθεση της συναδέλφου Λάτφορτ και αναμένω όπως είπα την προσαρμογή της. Γιατί δεν είναι δυνατόν να εκδίδονται εντάλματα σύλληψης για το ότι κάποιος δεν επέστρεψε έγκαιρα τη βιντεοκασέτα. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου αυτά, έχουν συμβεί. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κέρκοπ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι το ένταλμα σύλληψη όπω και το ένταλμα έρευνα ή εντολή έρευνα τέλο πάντων είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά για τα σοβαρά δικήματα και για την τρομοκρατία. Συγχαρητήρια στου εισηγητά. Η χώρα μου ωφελήθηκε από το ένταλμα σε πολλέ περιστάσει για την έκδοση κάποιων ε, βιβλιαστών, λαθρεμπόρων, τρομοκρατών ε, ε, παιδεραστών και θυμάμαι ότι παλιότερα τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα, υπήρχαν πολιτικά προβλήματα, περιπλοκές, γραφειοκρατία. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε τις μέρες εκείνες, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που η τρομοκρατία και το έγκλημα μας απειλεί κάθε μέρα. Και οπότε είναι ξεκάθαρο το σημερινό κόσμο ότι χρειάζονται αποτελεσματικά μέτρα, έγκαιρα μέτρα όσον αφορά την έκδοση των εγκληματιών. Πολύ σημαντικό, αλλά να υπάρχουν επομένω βέβαια και κάποιες, ε, κάποια, κάποια αντίβαρα ε, και να υπάρχει αναλογικότητα. Το έντομα σύλληψη προβλέπει ε, το ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη προφυλάκηση και έχουμε επομένω. δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ελαφρά εγκλήματα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, σύμφωνοι, είναι εξαιρέσεις αυτές οι, αυτές αλλά και αυτή η κατάχρηση είναι απαράδεκτη. Οπότε θα πρέπει να γίνουν κάποιες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Θέλουμε να υπάρχει δίκαιη δίκαιη, να υπάρχει αναλογικότητα και θα πρέπει οι εγκληματίες να μην μπορούν να κρυφθούν πουθενά στην Ένωση. Θα πρέπει όμως να καταπολεμούμε το έγκλημα μέσω του να υπάρχει πεποίθηση δικαίου στον κόσμο να υπάρχει εμπιστοσύνη στο σύστημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από όλα, πάνω απ' όλα, να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Πέτυχαν μια έξοχη τεκμηριωμένη έκθεση και βελτιώνει αυτό το αντικατάστατο εργαλείο για την αντιμετώπιση του συνοριακού εγκλήματος στην Ευρώπη. Η έκθεση αποκαλύπτει κάποια κενά όσον αφορά τη λειτουργία του μέσου αυτού και αυτό αποδεικνύεται και με στατιστικά στοιχεία. Από το 2005 μέχρι το 2009 μόνο το 1 πέμπτο των ενταλμάτων εξετελέστησαν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα και μειονεκτήματα θα πρέπει να προτείνουμε συνεπώς βελτιώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιφορτιστεί με τις σχετικές ε, προτάσεις. Είμαι σίγουρος ότι το νομικό πλαίσιο του κανονισμού είναι κάπως αόριστο και τα κράτη-μέλη μπορούν να δρούν κατά το δοκούν. Εάν βελτιώσουμε το σύστημα, τότε το ποσοστό των εκτελέσεων των εντολών θα αυξηθεί και αυτό. Ευχαριστώ. Ο κ. Μπάτεν έχει το λόγο. Ακούμε πολλά για θεμελιώδη δικαιώματα εδώ πέρα. Στην Αγγλία είχαμε πολύ καλά θεμελιώδη δικαιώματα πολύ πριν προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαν επί σειρά αιώνων με το Χάμπιος Κόρπους ε, καταρτιστεί το δικαίωμα δικαιωμάτων, η και ότι πρέπει να αποδειχθεί η ενοχή, ο καθένα θεωρείται ε, αθώος μέχρι αποδείξει των αντίου, όλα αυτά καταστρέφονται διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί το δικό τη σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη ήταν το αίτιο πολυάριθμων υποθέσεων πολλών αδικιών και θα αυξάνονται αυτέ οι περιπτώσει. Τώρα έχουμε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα έρευνα που θα δώσει δυνατότητα σε ξένε δυνάμεις να πετούν από να διενεργούν έρευνε εκ μέρου του και αυτό τότε θα έχουμε το προνόμιο να το πληρώνουμε. Η συμμαχία έχει την δυνατότητα να αυτοεξαιρεθεί από τα 135 μέτρα τη ποινική δικαιοσύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ανακοίνωσε ότι θα αυτοεξαιρεθεί από 100, αλλά θα συμμετέχει στα 35. 100 από τα οποία κάνουμε opt-out περιτεύουν ή ξεπερνιόνται από πιο πρόσφατη νομοθεσία. Τα 35 μέτρα όμως που επιλέγουν να συμμετάσχουν είναι τα χειρότερα και τα πλέον επικίνδυνα συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψης. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αναγκαίο, διότι ήδη υπάρχουν μέτρα αμοιβαία αρρωγή που επιτρέπουν στις αστυνομικέ δυνάμεις και στα δικαστικά συστήματα να συνεργάζονται μεταξύ του ε, σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό δεν αφορά συνεργασία, αφορά εναρμόνιση των νομικών μας συστημάτων επιδιώκοντας την μεγάλη ιδεολογική επίτευξη. Να πετύχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες της Ευρώπης. Αν ο Ντέβιτ Κάμερον είναι σοβαρός, περί επαναπατισμού των εξουσιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη χρυσή ευκαιρία να το κάνει αυτό τώρα. Υπάρχει ακόμα χρόνο να αλλάξει η απόφαση και να αυτοεξαιρεθεί η Βρετανία από όλα αυτά τα μέτρα προστατεύοντα τα πραγματικά συμφέροντα και ελευθερίε του Βρετανικού λαού. Φοβάμαι όμω ότι στην Δυτική θα κάνουν αυτό που έκαναν πάντα και θα απολύσουν του συμπολίτε του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενη Ομιλήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, Συμφωνώ απολύτω ε, με την ε, Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα. Ε, τι ακριβώ είναι, δίνει τη δυνατότητα σε ένα κράτο μέλο να ζητήσει από άλλο κράτο μέλο να κάνει κάποιε έρευνε για να λυθούν ε, περιπτώσεις σοβαρού εγκλήματος, ε, εμπορίας ανθρώπων, ε, παιδικής πορνογραφίας, διακίνησης ναρκωτικών. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαζόμαστε στενά. Το έγκλημα γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο και κινείται όλο και περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα στις αρχές να πιάνουν τους εγκληματίες όταν κινούνται διασυνοριακά το θέμα είναι η αναγνώριση των δράσεων άλλων κρατών μελών και ε, να βοηθάμε ένας τον άλλον ε, στις έρευνες. Οι εθνικές ε, αρμοδιότητες γίνονται απόλυτα σεβαστές και θα συνεχίσει να ισχύει το εθνικό ποινικό δίκαιο της κάθε χώρας. Ε, απλοποιούνται οι κανόνες αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Θα είναι πιο ε, εύκολο να εργάζονται αποτελεσματικά. Ε, για παράδειγμα, η εισαγωγή σαφών προθεσμιών θα επιταχύνει τη συλλογή σημαντικών στοιχείων από άλλο κράτος μέλος. Επίσης, είναι σημαντικό να εισάγουμε σαφή εχέγγυα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υπόπτων και να έχουμε και σαφείς κανόνες περί προσφυγών. Κύριε Πρόεδρε, η αυξημένη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική καταπολέμηση του διασυνοριακού εκκλήματος. Ε, το, η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας μαζί με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ε, αποτελούν πολύ καλά παραδείγματα του τι μπορούμε να κάνουμε μαζί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο να ωφελεί στην πραγματικότητα τους Ευρωπαίους πολίτες. Με ε, την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας μπορούμε να αυξήσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας ε, σεβούμενη ε, παράλληλα και την ε, ακαιρεότητα. Είναι λοιπόν σημαντικό βήμα για να δημιουργήσουμε μια περιοχή ελευθερίας και ασφάλειας στην Ευρώπη όπως ζητά το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τρία λεπτά συνάδελφος Βάιντεν Χόλσερ. Σας ευχαριστώ. Με το, την ε, Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας έχουμε ένα σημαντικό μέσο ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία. αυτό είναι απαραίτητο για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι η πρωτοβουλία αυτή προέρχεται όχι από την Κομισιόν αλλά από κράτη-μέλη μεταξύ άλλων την Αυστρία δείχνει ακριβώς ότι ε, τα εθνικά συμφέροντα δεν αντίκεινται στα ευρωπαϊκά. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε προσθέμενη αξία στον τομέα της ε, πολιτικής ασφαλείας. Έτσι θα διευκολυνθεί η ποινική δίωξη ε, στην Ευρώπη και θα εξαλειφθούν κάποια εμπόδια. Η Ευρωπαϊκή Εντολή έρευνας θα επιταχύνει τις διαδικασίες και θα τις κάνει πιο αποτελεσματικές. Ποιος μπορεί να είναι εναντίον. Η αξία ενός τέτοιου μέσου δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Συχνά υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία δυσκολεύουν ή εμποδίζουν τις αστυνομικές έρευνες. Αυτό λοιπόν δεν είναι προς όφελος των πολιτών που έχουν δικαίωμα στην προσωπική ασφάλεια. Ταυτόχρονα θα πρέπει να Γνωρίζουμε ότι ο, ο τομέας της ποινική δίωξης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και θα πρέπει να προσέξουμε να ε, προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των υπόπτων. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και η θέσπιση τους ε, στη συνθήκη είναι θεμελιώδη σημασίας και χαίρομαι πάρα πολύ που στις ε, διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο ήταν δυνατόν στο άρθρο 10 να έχουμε μια ρήτρα περί θεμελιωτών δικαιωμάτων. Ε, μια ευρωπαϊκή εντολή έρευνας μπορεί να ε, εκδοθεί εφόσον δεν θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα του υπόπτου. Επίσης, στο άρθρο 5 διασφαλίζεται να χρησιμοποιούνται μόνο μέτρα τα οποία επιτρέπονται στο κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας έτσι ε, περιορίζεται ε, σημαντικά και αποτελεί ε, μια επιτυχημένη προσπάθεια να αποφευθούν οι καταχρήσεις. Το Κοινοβούλιο με τις τροπολογίες του δείχνει ότι η προστασία των θεμελιωτών δικαιωμάτων και η ενισχυμένη αστυνομική συνεργασία στην Ευρώπη είναι συμβατά μεταξύ τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θέρμα τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για την καλή και εντατική συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βοητσεκόφσκι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το, η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα είναι πολύ σημαντική απόφαση και η έμπρακτη της ε, ε, ε, εφαρμογή και σημασία θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το Ευρω... αυτή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ε, Σύλληψης γιατί θα καλύψει πολύ περισσότερες περιπτώσεις, διασυνοριακές περιπτώσεις, ακρόαση μαρτύρων, αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων σε άλλο κράτος μέλος, οπότε σίγουρα οι αρχές επιβολής τάξης θα και του νόμου θα χρησιμοποιήσουν ιδιαίτερα αυτό το μέσο, την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. Επίσης ε, θα ήθελα να πω ότι η σύσφυξη της συνεργασίας ε, μεταξύ των δικαστικών αρχών ε, είναι πολύ σημαντικό θέμα, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το επίπεδο της απονομής δικαιοσύνης στα κράτη-μέλη, γιατί πολύ συχνά οι πολίτες παραπονιούνται για την απονομή της δικαιοσύνης. Θα πρέπει λοιπόν Πρώτα να εξασφαλίσουμε ότι η απονομή της δικαιοσύνης και ο δικαστικός κλάδος ε, χαίρει της εμπιστοσύνης των πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπονανίνη έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τη ευρωπαϊκή αυτή εντολή έρευνας και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι θέματα κλειδιά για να δημιουργηθεί ένα χώρο ποινικού δικαίου στην Ευρώπη. Η έκθεση του συναδέλφου Μέλλον εισάγει ε, μέτρα καταπολέμηση τη εγκληματικότητα πιο αποτελεσματικά από αυτά προσφέρει η δικαστική παραδοσιακή συνεργασία. Ταυτόχρονα, η ανάγκη να εξασφαλίζεται ο σεβασμό των θεμελιών δικαιωμάτων του ανθρώπου που εκφράζονται στην ε, συνθήκη όσον αφορά τι έρευνε είναι ένα στόχο προ επιδίωξη και πρέπει να κινηθούν προ την κατεύθυνση και οι διατάξει του άρθρου 5 και 6 σχετικά με αυτό είναι κάτι που στηριχθεί. Ο έλεγχο που γίνεται για την εφαρμογή του εντάλματο σύλληψη έδειξε σημαντικέ τρευλώσει όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου και πώ χρησιμοποιήθηκε από τα διάφορα κράτη-μέλη το μέσο. Και υπάρχουν και διάφορα κενά τη νομοθεσία που κάνουν αβεβαιότητα, την προστασία, αβεβαιότητα, δίνουν αβεβαιότητα στην προστασία ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 τη Χάρτη των Δικαιωμάτων θα πρέπει η αρχή που εκδίδει ένα ευρωπαϊκό ένταλμα να μπορεί να ελέγχει την αλογικότητα του μέτρου θα πρέπει ε, να, μην, να αποφεύγεται η μη χρησιμοποιημένη ε, ισορροπημένη χρήση του εντάλματος. Θα πρέπει να προστατεύονται λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρομαι στην υποχρέωση που έχουν τα κράτη-μέλη να εγγυώνται το δικαίωμα σε προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 13 των Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά την εκτέλεση ενό μέσου το οποίο υπόκειται στο πλαίσιο αμοιβέ αναγνώριση. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γιακολίνο έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Προέδρε, κυρία Επίτροπε Ρέντινγκ. Αναμφισβήτητα τα δικαστικά μέτρα που σήμερα συζητούμε είναι αδιαμφισβήτητα σημαντικά για την οικοδόμηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης και στο ποινικό τομέα. Αλλά αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης περνούν από μέσα που έχουν σημαντικούς στόχους και γι' αυτό χρειάζεται και αμοιβαία αναγνώριση και ταχεία εκτέλεση από τα κάτι μέλη των μέσων αυτών. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συλλήψης είναι η σωστή σκέψη που εξεφράστη από, τον, από την εισηγήτρια Ράτφορντ όσον αφορά την χρήση σύμφωνα με κριτήρια αυστηρής αναλογικότητας, διότι χρειάζεται να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα από τη μια και από την άλλη πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα όσον αφορά την καταπολέμηση και την εξυχνίαση κάποιου κλίματο. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο Μέλο για την έξοχη δραστηριότητα του όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εντολή Απόδειξης Λοιπόν, το, θα πρέπει ε, να υπάρχει βεβαιότητα, διότι πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις για να εκδίδεται αυτή η εντολή. Ε, η δικαστική συνεργασία και η αστυνομική συνεργασία είναι ουσιαδιώδη στοιχεία για να δημιουργηθεί ο χώρος δικαιοσύνης, ούτως ώστε να το, για το πετύχουμε αυτό πρέπει να μειώσουμε προφανώς την χρήση του εντάλματος, του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ε, περίπτωση υπερεθνικού εγκλήματος και όπου χρειάζεται η προσφυγή σε μέτρων που προσωρινής κράτης. Όσον αφορά το ευρωπαϊκή, την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας, θα πρέπει το κόστος να το φέρει το κράτος εκτέλεσης. Και θα πρέπει να αναγνωρίζεται και ακρόση των μαρτύρων και μέσω βιντεοδιασκέψεων. Σίγουρα το σύστημα της πληροφορικής είναι ένα μοντέλο αναφοράς και σε οργανωτικό επίπεδο. Και τέλος κλείνω λέγοντας κυρία Πρόεδρε ότι είναι σημαντικά αυτά τα μέσα και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην επόμενη Ολομέλεια του Μαρτίου θα εξετάσουμε προκαταρκτική έκταση που ελπίζουμε να προσανατολίσει μελλοντικής, ε, τις μελλοντικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μωράς έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ε, ε, Πρόεδρε, πριν λίγους μήνες υπέβαλα στοιχεία στη Βουλή των Λόρδων σχετικά με την αποτελεσματικότητα ε, του, της Ευρωπαϊκής Ενταλής Έρευνας και κατά τις έρευνές μου ε, έμαθα ότι ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό μέσο, ότι αποτελεί θεμελιώδη λίθο της διασυνοριακής συνεργασίας. Όπως όμως όλοι γνωρίζουν, ε, απαιτεί το και άμεση και σαφής μεταρρύθμιση. Οι εργασίε τη Βαρόνη Λάτφορντ ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικέ και η ομάδα μα πολύ ευχαρίστω θα τι υποστηρίξει. Ε, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα ε, του πόσο κακή είναι η διασυνοριακή συνεργασία. Πρέπει όμως ε, να έχουμε σαφή στοιχεία σχετικά με το τι έχει πάει στραβά. Στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε την περίπτωση ε, της ε, Μάγκη Χιούς και του ε, γιου της Ρόμπερτ που, στους οποίους επιτέθηκαν όταν βρίσκονταν σε διακοπές στην Κρήτη. Έγινε η σύλληψη των ε, ενόχων. Ε, επίσης, ε, λόγω του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης συλλήφθηκαν οι ένοχοι για τις βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο το 2005. Υπάρχει όμως, υπάρχουν περιπτώσεις υπερβολικού χρόνου προφυλάκησης. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε την σωστή ισορροπία και με τρόπο αντικειμενικό και ισορροπημένο να εφαρμόσουμε την μεταρρύθμιση. Α κάνουμε τη δουλειά μα δηλαδή για να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση, αλλά όταν εργαζόμαστε πάνω όταν εργαστήκαμε πάνω στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ε, διαπιστώσαμε κάτι ιδιαίτερα πολύτιμο. Ότι εδώ στη διασυνοριακή δικαιοσύνη κάνουμε κάτι πολύ αποτελεσματικό για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει όμως να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Μωράες, υπάρχει γαλάζια κάρτα για σας. Okay. Please. Claude, can I ask you to... Κλοντ, να σου επιτρέψω να, να, ε, να μου επιτρέψεις να σου ζητήσω να ανακαλέσεις κάτι. αναφέρθηκε ε, στην κυρία Χιούς ε, και είπες ότι δικάζονται όσοι του επιτέθηκαν. Όχι, όσοι κατηγορήθηκαν ότι επιτέθηκαν. Κάποιοι έχουν αποδείξει ότι δεν ήταν καν παρόντες κατά την στιγμή της επίθεσης. Ωστόσο, η έλλειψη στοιχείων δεν έχει εμποδίσει την έκδοση τους. ξέρω ότι είσαι πολύ δίκαιος ε, άνθρωπος. Μήπως θα ήθελες να ανακαλέσεις τη λέξη ε, αυτή που επιτέθηκαν και να πεις ε, οι κατηγορούμενοι. Ναι. Θα έπρεπε να διαβάσω την ομιλία μου. είπα λοιπόν ότι όσοι επιτέθηκαν ε, δικάζονται, αλλά νομίζω ότι έχεις δίκιο. Μάλλον δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα, αλλά ναι, νομίζω ότι έχεις δίκιο. Ε, κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν μου έχουν δώσει γαλάζια κάρτα. Επιτρέψτε μου ε, να εξηγήσω στον συνάδελφο ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα ε, γρήγορη δίωξη ε, ανθρώπων λόγω του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη. Ξέρω ότι έχει παραδείγματα περιπτώσεων που πήγαν στραβά. Ε, Ακριβώ γι' αυτό θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη και ελπίζω να το σεβαστεί αυτό. Σας ευχαριστώ, κύριος Νίκολσον, για ένα λεπτό. Uh, ευχαριστώ. Εγώ κατάγομαι από τη Βόρεια Ιρλανδία και εμείς είμαστε το μόνο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει ε, σύνορο με άλλο κράτο Και μάλιστα τα σύνορα αυτά ε, υποτίθεται ότι ε, ήταν ε, δύσκολα και δύσκολη αντιμετώπιση τη διασυνοριακή συνεργασία. Χρειάζεται πολύ στενή διασυνοριακή συνεργασία και αστυνομική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματο. Και θα ήθελα να απαντήσω φόρο τιμή ε, στι αστυνομικέ δυνάμει τη Βορείου Ιρλανδία ε, για τον τρόπο με τον οποίο εφάρμοσαν αυτή την αστυνομική συνεργασία που στο παρελθόν δεν υπήρχε καν. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχουμε για την καταπολέμηση της διασυνοριακής τρομοκρατίας. Χωρίς αυτό το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης δεν θα είχαμε νόμιμη, βάση για έκδοση ε, ε, μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Βορείου Ιρλανδίας. Χρειαζόταν λοιπόν κάτι τέτοιο και χρειαζόμαστε έντονη αστυνομική και δικαστική συνεργασία γιατί μια έλλειψη τέτοια συνεργασίας θα ευνοήσει μόνο τους τρομοκράτες και τους εγκληματίες. Και μάλιστα μεταξύ το 2004 και το 2013 είχαμε σύλληψη πολλών τέτοιων υπόπτων. Βέβαια θα πρέπει να εφαρμόσουμε και την αρχή της αναλογικότητας. Πάντως ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια γιατί θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψη έχει πολύ μεγάλα πλέον εκτήματα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Στίερ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ είμαι υπέρ της ενίσχυσης ε, του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως ε, για το ποινικό δίκαιο, για τα ποινικά θέματα και θεωρώ ότι η σχετική οδηγία αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί θα διευκολύνει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τα εγκλήματα που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Επίσης, ε, θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη εξακολουθεί να είναι ο πιο επιτυχημένο μηχανισμό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποινικό δίκαιο. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα βελτίωση ε, με ε, την ε, αποφυγή πρώτα απ' όλα πολιτικής επιρροής σε ό,τι αφορά τις αιτήσει για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Σίγουρα η απόφαση για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τη διαδικασία έκδοσης ή να, υπο, επιβαρύνεται με πολλές γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Σε καμία περίπτωση πάντως θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης να γίνει αντικείμενο πολιτικής χειραγώγησης. Είχαμε στην περίπτωση της Κροατίας ένα τέτοιο αίτημα για ένα πρώην ε, υπάλληλο της ε, ε, των μυστικών υπηρεσιών και δείχνουν ότι οι πολιτικές τέτοιες δομές είναι ακόμη ισχυρές και μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εξουσία τους για χειραγώγηση για της κοινή γνώμη και για άσκηση επιρροής και στη δικαιοσύνη. Εμείς καταφέραμε ε, να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση και χάρη στην άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι απο, ήρθαν τα εμπόδια για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ε, και δόθηκε ευκαιρία στους δικαστές και όχι στους πολιτικούς για να αποφασίζουν για την τύχη ε, πρώην, ε, μελών του, των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό ήταν πολύ θετικό, πολύ θετικό βήμα γιατί μερικοί ε, αφισβήτησαν την ικανότητα της Κροατίας να εφαρμόσει από την 1η Πρώτου ε, του 2014 13 ε, καθήκοντά της. Σε κανένας δεν θα πρέπει να εκφεύγει του νόμου. Αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον μας, γιατί δεν νοείται οικονομική και κοινωνική πρόοδος χωρίς το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν είναι στην αίθουσα η κυρία Φρασίκοβα. Μπένοβα. Δίνω το λόγο για την προσέγγιση προσοχής του Προέδρου στην συνάδελφο Μορκουνάιτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να πω μερικά λόγια όσον αφορά το θέμα που συζητάμε και θα ήθελα να πω και τις απόψεις μου για τη θέση της ηγήτριας. Πρέπει να εφαρμόζουν τα ίδια μέτρα τα κάτι μελη όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα ε, κάποια χώρα κάποτε είχε αρνηθεί να εκδώσει κάποιον που ήταν ύποπτος για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και για εγκλήματα πολέμου επικαλούμενοι διαδικαστικά επιχειρήματα. Το 1991, 13 Ιανουαρίου, αυτό το άτομο διέπραξε όμως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λιθουανία και δεν μπόρεσε να εκδοθεί αυτό το άτομο στη Λιθουανία. Δεν μιλάμε στην έκθεση για ενδεχόμενες εξαιρέσεις σύμφωνα με τις οποίες για την έκδοση του εντάλματος σύλληψη εγκλήματα που διαπράχθηκαν μετά το 2000. Αυτή η εξαίρεση δεν θα πρέπει να ισχύει για εγκλήματα κατά ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που είναι πιο σοβαρά. Και δεν υπάρχει παραγραφή αυτών στο διεθνέ δίκαιο. Έχει κάνει η πρόταση σχετική Ευρωπαϊκή Πίτρο στο κρατη Η Κροατία και τα νέα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να μην το εφαρμόσουν αυτό θα ήθελα να ζητήσω κάποια διευκρίνηση από την Επίτροπο Ρέντινγκ. Τι σκεφτόσαστε όσον αφορά την παραγραφή εγκλημάτων και τη δυνατότητα να εφαρμόζονται αυτό το Ευρωπαϊκό Έντομα και η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα για εγκλήματα που διαπράχθηκαν μετά το 2000. Ευχαριστώ, Τόμασίτ, συνάδελφο Τόμασίτ. Ή συνάδελφο. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη είναι σημαντικό εργαλείο για τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, διότι θέτει τέρμα στην καριέρα εγκληματιών που κρυβόταν και κρυβόταν λόγω κακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών. Για την Κροατία αυτό είναι κάτι σημαντικό διότι οι πολίτες της ήταν θύματα συστηματικής δίωξης από τι Ιουγκοσλαβικέ μυστικές υπηρεσίες. Θα ήθελα να καλωσορίσω ιδιαίτερα αυτό το ψηφισμά εκεί που καλεί για συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση των ειδικών νομικών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Στην Κροατία ένα δικαστήριο αποφάσισε να εκδώσει τον κύριο Πέκοβιτ στη Γερμανία λόγω του φόνου Κροάτου μετανάστη. Ένα άλλο δικαστήριο όμως δεν εξέδωσε ένα άλλο άτομο που περιελβαλανόταν στο ίδιο ένταλμα. Και γι' αυτό φαίνεται πόσο σημαντικό είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ο συνάδελφος Μπίελαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη ε, στόχο έχει την επίσπευση των ε, διαδικασιών για την άμεση παραπομπή υπόπτων και κατηγορουμένων στα δικαστήρια καταργήθηκαν ε, κάποιες ε, διοικητικές φάσεις ε, για την λήψη των αποφάσεων, κάτι που περιόρισε σημαντικά τον χρόνο της έκδοσης. Σε μια κατάσταση ανοιχτών συνόρων, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μηχανισμού και να μηχανισμούς και να εξασφαλίζουν την προσαγωγή των εγκληματιών στη δικαιοσύνη. Φυσικά υπάρχουν κάποιες ατέλειες στο σύστημα αυτό για παράδειγμα, η υποτιθέμενη επιλεκτικότητα των δραστηριοτήτων των αρμοδίων αρχών που οδηγεί μερικέ φορές σε κατάχρηση του μηχανισμού αυτού ή σε μη εφαρμογή τη αρχή τη αναλογικότητα. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για σύσφυξη τη συνεργασία προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη και σε καμία περίπτωση να μην κλονιστεί η αξιοπιστία του. Συνάδελφε Πάσκα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ο ευρωπαϊκός αυτός χώρος που θέλουμε να δημιουργήσουμε απαιτεί καθορισμό της αποτελεσματικής συνεργασίας των δυνάμων ασφαλείας και των δικαστικών αρχών όταν διώκουν διασυνοριακούς εγκληματίες. Το, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Ένταμα του 2002 δημιουργεί την αναγκαιότητα να αναγνωρίζονται οι διάφορε διαδικασίε των κρατών μελών, να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει διάφορα κενά και λήψει όσον αφορά τη λειτουργία των υφισταμένων συστημάτων. Άρα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει, να προτείνει κάποια νομοθετικά μέτρα για να καλυφθούν τα κενά. Θα πρέπει πέρα από τα πορίσματα που παρουσιάζονται στην έκθεσή της, να διενεργήσει μια ανάλυση της μη εκτελέσεως των ευρωπαϊκών ενταλμάτων συλλήψεως για να εντοπιστούν οι τομείς εκεί που δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος η κυρία Ρέντινγκ έχει τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους αξιότιμους ευρωβουλευτές ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες στους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων που διαφέρουν από τους κανόνες που ισχύουν σε άλλους πολιτικούς τομείς. Για παράδειγμα, με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας, τα κράτη-μέλη δίνονται να υποβάλουν ε, νομικές προτάσεις χωρίς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ισχύει για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα, για παράδειγμα. Ευτυχώ στην περίπτωση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί τη διαδικασία με βάση τη διαδικασία συναπόφαση και θα υποβάλει προτάσει που θα εξισορροπήσουν ε, το στόχο τη ασφάλεια με το στόχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πριν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα, τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να υποβάλουν ε, προτάσει ε, τα κράτη-μέλη χωρί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χωρί έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευτυχώς ε, η κατάσταση αυτή σταματά από την 1η Δεκεμβρίου και θα ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση εξαίρεσης χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό, την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα, θα ήθελα να πω ότι ευελπιστώ ότι η οδηγία αυτή θα εφαρμοστεί αυτή τη φορά και δεν θα ισχύσει αυτό που συνέβη με το πλαίσιο για την εντολή συλλογή αποδείξεων που εφαρμόστηκε μόνο από δύο κράτη-μέλη. Θα ήθελα επίσης να πω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η εφαρμογή τη οδηγία αυτής μπορεί να παρακολουθηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα διστάσει να ξεκινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων για ελλειπή σωμάτωση στην εθνική νομοθεσία ή ε, μη εφαρμογή των κανόνων. Το ίδιο ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, γιατί από την 1η 12 η μεταβατική φάση που προβλέπει, η μεταβατική περίοδος που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας ολοκληρώνεται και από την 1η Δεκεμβρίου και μετά θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει κυρώσεις για την ελλειπή ή ατελή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Στόχος μας είναι η πλήρης εφαρμογή και από αυτή την άποψη ε, μηχανισμοί όπως ε, η Ευρωπαϊκή Εντολή Εποπτείας Επιτήρησης ε, επιτρέπει να περιορίσουμε τους χρόνους προφυλάκηση σε υποθέσεις του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψη. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλα τα εργαλεία που θα πρέπει να λειτουργούν ε, από κοινού και εύρυθμα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι εδώ και πολλά χρόνια καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια και ήταν πολύ σημαντικό έργο. Για παράδειγμα, τα δικαιώματα της δίκαιης δίκης είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα για να εξισορροπηθεί ο στόχο τη ασφάλεια με τον στόχο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των πολιτών. Όλε αυτέ οι κατευθυντήριε γραμμέ και οδηγίε περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία που ενισχύουν την εφαρμογή του εντάλματο σύλληψη. Δικαίωμα σε μετάφραση και διερμηνία. Δικαίωμα σε ενημέρωση για τα δικαιώματα. Δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο. Ακόμη ε, και στη ε, δικηγόρο στη χώρα προέλευσης και στη χώρα προορισμού του εντάλματος σύλληψης. Όλα αυτά τα δικαιώματα πλέον κατοχυρώνονται. Ε, δικαίωμα ευεργέτημα παινίας, τεκμήριο αθωότητας, δικονομικά δικαιώματα ανηλίκων και ευάλωτων ατόμων. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για να εξασφαλιστεί η ισορροπία που δυστυχώς δεν ίσχυε στην κατάσταση πριν τη συνθήκη της, πριν τη συνθήκη Τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει όλες αυτές τις αρχές. Και λυπούμε ειλικρινά που μερικά κράτη-μέλη αρνούνται τη συμμετοχή σε όλα αυτά τα στοιχεία των δικαιωμάτων της δίκαιης δίκης. Γιατί κάτι τέτοιο με τέτοια αυτοεξαίρεση δεν είναι καθόλου θετική για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Το λόγο έχει ο κύριος Μέλο για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, αυτό που θα μας επιτρέψει η οδηγία είναι περισσότερη δικαιοσύνη, γιατί θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ε, ποινικών ε, ερευνών, μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας. Ο κύριος Μπάτεν εξανέστη γιατί είπε ότι οι αστυνομικοί θα πρέπει, οι Ευρωπαίοι αστυνομικοί θα πρέπει να διαρευνήσουν ε, εγκλήματα. Μα φυσικά και θα πρέπει να διαρευνήσουν εγκλήματα. Επίσης εξανέστη γιατί ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ξοδέψει κάποια χρήματα. Φυσικά και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία και η Πορτογαλία και η Ισπανία, όλες οι 28 ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αφιερώσουν κάποια κονδύλια. Αλλά είναι μια προτεραιότητα ε, που μας ε, επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός ε, Κοινός Χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει ο όποιο διαπρέπει το έγκλημα να γνωρίζει ότι το έγκλημά του δεν θα μείνει ατιμόρυτο. θα δικαστεί σε αμερόληπτο δικαστήριο και μάλιστα με συγκέντρωση συγκεκριμένων αποδείξεων. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία, ο ύποπτο θα αθωωθεί. Και όλα αυτά είναι, γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένα χώρο ελευθερία. Γιατί Κάθε μέρα καθιερώνουμε αυτή την ε, ελευθερία και επίσης ε, κατοχυρώνουμε όλους τους μηχανισμούς, τα εργαλεία και τις ε, δικονομικές και ουσιαστικές εγγυήσεις ενός κράτους δικαίου. κατοχυρώνονται αυτές οι εγγυήσεις για όλους, και για τους υπόπτους και για τους κατηγορούμενους. Πρέπει όμως να έχουμε μία βεβαιότητα ότι από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ ο χώρος Σέγγεν και επέτρεψε την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, σίγουρα με αυτήν την ελεύθερη διακίνηση διαπράττονται και πιο εύκολα εγκλήματα. Και θα η δικαιοσύνη των χωρών θα πρέπει να παρακολουθήσει αυτές τις ε, ροές και θα πρέπει να μπορεί να δώσει απάντηση στα προβλήματα. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα έχουμε ένα ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, γιατί θα έχουμε αποτύχει στον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να ευχαριστήσω θερμά τους και τους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λάτφορντ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνο με ε, σχεδόν όλους όσους μίλησαν και τους ε, ευχαριστώ θέρμα που συμμετείχαν. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ ιδιαίτερα στις ε, παρατηρήσεις του κυρίου Νίκολσον σχετικά με την κατάσταση στην Ιρλανδία. Συμφωνώ ακόμα και με τον Πάτεν σχετικά με το ότι πρόκειται για κατηγορούμενους και όχι ενόχους δεν ε, θα εκπλήξει όμως τον κύριο Μπάτεν ότι κατά τα άλλα διαφωνούμε και εγώ θα ε, χαρώ πολύ να δω την, ε, την μονομαχία μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη διάρκεια της προφυλάκησης και τις κακές συνθήκες φυλάκησης. Αυτό είναι κάτι που υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και καλούμε την Επιτροπή να εξερευνήσει όλους τους διαθέσιμους τρόπους για να βελτιωθεί η κατάσταση. Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω, ε, επειδή αναφέρθηκε η καλύτερη κατάρτιση από κάποιον, είναι η καλύτερη κατάρτιση των ε, επαγγελματιών ε, στον τομέα του δικαστικού και των ε, δικηγόρων υπεράσπισης. Συμφωνώ όμως απόλυτα με την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ σχετικά με την σημασία της οδηγίας για τα δικονομικά δικαιώματα. Πιέζω την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διότι θέλω να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Εντολή Εποπτείας. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που ε, έχει επιλέξει να συμμετάσχει στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που η έκθεσή μου καλεί να γίνει γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή των μέσων που υπάρχουν, μεταξύ άλλων της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας. Όμως απογοητεύτηκα κάπως με την έλλειψη μιας προορατικής ε, αντιμετώπισης από την κυρία Ρέντινγκ. Είπε ότι οποιοδήποτε άνοιγμα της συζήτησης για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα θα ήταν κάτι πρόημο αυτή τη στιγμή. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε αρκετό υλικό στη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Θα ήθελα λοιπόν να ασκήσω πίεση στην Κομισιόν και προσβλέπω στην καλή συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν για να λάβουμε μέσα στην ε, επόμενη χρονιά πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσατε τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν επιτρέπετε να την αγνοήσετε. Um, Υπάρχει γαλάζια κάρτα για σας. Mr. Button. Ο κύριος Μπάτεν. Ευχαριστώ. Σάρα, μίλησες για υπερβολική διάρκεια της προσωρινής κράτησης και θα πρέπει να αποφεύγεται, συμφωνώ. Ένας από τους λόγους γι' αυτό είναι ότι όταν εκδίδονται κάποιοι στη Βρετανία, η αστυνομία θα πρέπει να είναι έτοιμη για την υπόθεση. Πρέπει να ετοιμάσει ε, τη δικογραφία πριν να εκδοθεί κάποιο Στην υπηρετική Ευρώπη υπάρχουν κάποια συστήματα όπου οι ε, εισαγγελίε που διενεργούν την έρευνα μπορεί να χρειαστούν μήνε και χρόνια για την έρευνα και αυτοί κρατούνται το μεταξύ. Κάθε αστυνομική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ετοιμαστεί ε, πλήρω όσον αφορά την υπόθεση και την δικογραφία που ζητήσουν να παραδοθεί ένα ε, που πρέπει να δικαστεί. Συμφωνώ μαζί σα, λέει κυρία Λάτφορντ. Ο τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη είναι ότι σε, πριν από τη δίκη υπάρχει κράτηση για λόγου ποινική δίωξη. Όχι για του λόγου έρευνα. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι το σημαντική Ευρωπαϊκή Εντελή Έρευνα. Για να φύγει κάποιο βάρο από το Ευρωπαϊκό Ένταλμο. Ένταλμα ε, σύλληψη. Χρειάζεται και διαβούλευση. Και θα είναι πολύ σημαντική. Τα δικαστήρια των χωρών θα μπορούν να διαβουλεύονται. Υπάρχουν διάφορα συστήματα στα κράτη-μέλη. Δεν, ε, δεν ε, θέλουμε να πετύχουμε όμορφο ποινικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή είναι η σημασία της αμοιβή αναγνώριση. Διότι αν είναι μακρά η προσωρινή κράτηση, αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Το είπα και υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έχουμε τον Άντιο Σίμιου που πέρασε φρικτή εμπειρία που δεν έπρεπε να του συμβεί διότι θα έπρεπε να αρνηθεί την έκδοση το Βρετανικό Δικαστήριο. Και είναι ψηφοφόρο μα. Το Ευρωπαϊκό Έντομα Σύλληψη πρέπει να χρησιμοποιείται για του σκοπού δίωξη. Όχι για να επιτυγχάνονται εκδόσεις για σκοπούς έρευνας. Σας ευχαριστώ. Η κοινή συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12.